Α μας. Ας φροντίσουμε λοιπόν να τις διεξαγάγουμε απρόσκοπτα. Η πρώτη έκθεση είναι της κυρίας Χαούταλα και αφορά την αίτηση άρση ασυλίας της κυρίας Μαρή, Μαρή Κριστίν Μπουτονέ. Συνήθις ψηφοφορία. Κανονικά ποιος είναι υπέρ της ε, αίτησης. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση Χαούταλα. Επόμενο θέμα είναι ο διορισμός του Σάιμον Μπουσούτιλ ως μέλους της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 255 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μυστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με σημαντική διαφορά. Επόμενο θέμα, η ονομαστική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες στην Ολομέλεια για την ονομαστική σύνθεση αυτής της Ειδικής Επιτροπής, οπότε χωρίς ε, τροπολογίες επιβεβαιώνουμε την ονομαστική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη έκθεση, τη σύσταση του κ. Μπορέλη για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισλανδίας για την προστασία γεωγραφικών ε, ενδείξεων, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση και πάλι του κυρίου Μπορέλη. Ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. έκθεση του κ. Χρυσόγονου με θέμα την εφαρμογή της οδηγίας για την διαμεσολάβηση. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση De Jong με θέμα τη λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Ο κύριος Ντε Γιόγκ, ο εισηγητής, ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ, έχετε δύο λεπτά. Παρακαλώ, κύριε Ντε έχετε το λόγο. Πατήστε και το κουμπί αν θέλετε. Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα μάλλον όχι, όχι κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν συζητήσαμε στην Ολομέλεια την έκθεσή μου, γι' αυτό θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει τις ε, συστάσεις ε, που έγιναν σχεδόν ομόφωνα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Οι εταιρείες συνήθως δεν πηγαίνουν, απευθύνονται στα δικαστήρια κατά των ε, μητρικών εταιριών τους, αλλά αυτά γίνονται όταν ε, γίνονται κατά χρήση του συστήματος ε, ή διόχρησης. Πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε η κατάσταση αυτή. Σας ευχαριστούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση ΚΡΕΛ για τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη. Και πάλι ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μίλαν Σβέρ για την πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξαποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη διαβίου μάθηση. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση της Καρή Μαντελή για την κατάργηση παροχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοείας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Και εδώ θα γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνατε. Έγινε δεκτή ε, η έκθεση της Καρή και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση. Έκθεση Ζωρίνια τώρα. Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες. Τροπολογία 30 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Διανατάσσεως της χειρός ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώνει και εδώ την πρώτη ανάγνωση στο θέμα αυτό. Έκθεση για Μπούζεκ για τα μέτρα κατοχήρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Τροπολογία 179. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 178. Κανονική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ, δυνατάσσος στις χειρός κατά αποχές εγκρίνεται και εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ανάγνωση επόμενο θέμα η φαλαινοθυρία στην Ορβηγία για διαδικαστικό ζητήσατε το λόγο όχι ωραία συνεχίζουμε τροπολογία 1 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο. Ποιος είναι υπέρ του αρχικού κειμένου. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ή μάλλον ε, διορθώνει ο πρόεδρος απορρίπτεται η τροπολογία 2 και μάλιστα με μεγάλη διαφορά οπότε ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της παραγράφου 2 ποιος είναι υπέρ του αρχικού κειμένου της παραγράφου 2 κατά αποχές εγκρίνεται το αρχικό κείμενο για την παράγραφο 2 με πολύ μεγάλη διαφορά και σας ζητώ συγγνώμη για το προηγούμενο λάθος μου. Τροπολογία 9 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά της τροπολογίας 9. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 9. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος ποιος είναι υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα για τη φαλαινοθυρία στην Ορβηγία Έκθεση Ρεβόντα Λόν και Κοράτσα Μπίλτ. Ο κύριος Γουλφ, διαδικαστικό. Ευχαριστώ. Με βάση το άρθρο 184, στο αγγλικό κείμενο, σελίδα 10 από 24, στο τμήμα 4, λέει ότι το Κοινοβούλιο τονίζει ιδιαίτερα ότι η άρνηση των, δικαιωμάτων, των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης έκτρωσης είναι βία κατά των γυναικών. Αυτή η ρήτρα μπορεί να κάνει όποιον θεωρεί ότι ε, ε, πρέπει να περιοριστούν οι εκτρώσεις, ότι είναι κατά των ε, εκτρώσεων να το κάνει να, είναι, ε, να υπόκειται σε ποινικό αδίκημα. Θα ήθελα οι νομομαθείς να εξετάσουν το κείμενο αυτό άλλη μια φορά, γιατί αλλιώ εκατομμύρια ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκληματίε αμέσω μετά αυτή την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Το σημειώνουμε. Περνάμε στην ψηφοφορία. Στην παράγραφο 4, τρία τμήματα, πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ. Αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, παράγραφο 4. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα του αρχικού κειμένου της παραγράφου 4. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για το τμήμα 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν χρειάζεται να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, είναι σίγουρο ότι εγκρίνεται. Παράγραφος 9 κάπα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, για το αρχικό κείμενο και πάλι, ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος 9 κάπα. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 4, εδάφιο M, σε δύο τμήματα για το αρχικό κείμενο και πάλι. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Αρχικό κείμενο. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο 15 αρχικό κείμενο τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται αλλά καλώς το ελέγξαμε τα μικρή διαφορά Αιτιολογική σκέψη 1 σε δύο τμήματα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματο, αρχικό κείμενο. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη R. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΑΑ, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, τι το άλλο είναι υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πολύ σημαντικό θέμα και συγχαρητήρια στις δύο συνεισηγήτριες. Έκθεση Μαρία Ρενά για το πρώτο 36 ε, ποιος είναι υπέρ σε δύο τμήματα κατά αποχές Ελεκτρονικός ηλεκτρονικός έλεγχος για το 46 πρώτο τμήμα του αρχικού κειμένου τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται δεύτερο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Περνάμε στις αιτιολογήσεις ψήφου.